και για το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2010. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι παρόντες στην αίθουσα και αρκετοί επίτροποι. Έχουμε λοιπόν πολυάριθμη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε υψηλότερο επίπεδο, κάτι που καταδεικνύει τη σπουδαιότητα αυτού του ζητήματος. Έχουμε λίγο περιορισμένο χρόνο εξαιτία τη ε, αναδιαμόρφωση τη ε, ημερήσια διάταξη. Μετά τη δήλωση του κυρίου Μπαρόζο, θα ακούσουμε του εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων που θα εκφέρουν την πολιτική γνώμη σε σχέση με τις προτάσεις του νομοθετικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2010. Και κατόπιν θα ξαναδώσουμε το λόγο στον κύριο Παρόζο, παρακαλώντας τον να σχολιάσει τις παρατηρήσεις των ε, αρχηγών των πολιτικών ε, ομάδων. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μπαρόζο. Σας ευχαριστούμε θερμά καταρχήν που ήρθατε και <laughs> μας επισκεφτήκατε. Για όλους μας ήταν δύσκολη η έλευση στο Στρασβούργο και ακόμη μερικοί δεν πρόλαβαν να φτάσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό και έχουμε τόσο μικρή προσέλευση. Αποφασίσαμε να αναβάλουμε και τι ψηφοφορίε σε αυτή την Ολομέλη, γιατί όλοι θα πρέπει να δίνονται να ψηφίζουν και ορισμένοι ευρωβουλευτέ δεν κατόρθωσαν καν να έρθουν στο Στρασβούργο. Έχουμε νέου κανόνε που ίσχυσαν για την παρούσα Ολομέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Έχω την τιμή και την ευχαρίστηση να σας παρουσιάσω το πρώτο πρόγραμμα εργασιών αυτής της Επιτροπής που αποτελεί και το πρώτο πρόγραμμα εργασίας από τη θέση ισχύ της Λισαβόνας. Έχω την τιμή και την χαρά να το πράξω την παρουσία όλου του επιτελείου μου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό προς δείγμα σεβασμού απέναντι στο Ευρωκοινοβούλιο. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν ε, το παρουσιάζουμε σε μια αποφασιστική ε, στιγμή για την Ευρώπη, διότι τώρα πρέπει να δράσουμε. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν προκύπτει από τον πολιτικό μας διάλογο μετά από έντονες διαβουλεύσεις ε, που στηρίχθηκαν τους πολιτικούς προσανατολισμούς που παρουσίασε για την προσεχή πενταετία το Κοινοβούλιο μου ανέθεσε τον Σεπτέμβριο την ευθύνη για μια δεύτερη εντολή. Μετά από τις ε, ακροάσεις οι οποίε επέτρεψαν να σφυριλατήσουμε μια κοινή άποψη σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, το Συλλογικό Όργανο των Επιτρόπων έλαβε την ψήφο εμπιστοσύνη σα τον Φεβρουάριο. Με άλλα λόγια, αυτό το πρόγραμμα εργασία καταδεικνύει μια σημαντική σύγκληση με τις πολιτικές επιθυμίες του σώματός σας. Προτελεί λοιπόν μια πλατφόρμα σταθερή για να πετύχουμε φιλόδοξα αποτελέσματα η πρώτη μας προτεραιότητα θα είναι ε, εξάρθουμε από την κρίση και να θέσουμε τις βάσεις για μια υφόρο ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Τα κατεπήγοντα ζητήματα. Συζητήσαμε τα τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του πρόσφατου ε, Συμβουλίου. Ο μηχανισμό λοιπόν για την υποστήριξη τη Ελλάδα, συστάθηκε στι 11 Απριλίου. Η Κομισιόν αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το μηχανισμό, ε, το οποίο θα θέσει σε ενέργεια όταν η Ελλάδα το ζητήσει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα για το ότι η Κομισιόν ευθύ εξ αρχή αναμίχθηκε για την εξέβρεση μια λύση στο δημοσιονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και στη διατήρηση της σταθερότητα εντό τη ευρωζώνη και αυτό το πράξαμε πάντα σεβόμενοι την αρχή της αλληλεγγύης αλλά και της υπευθυνότητα. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερο, να αναζητήσουμε γιατί προέκυψαν αυτά τα προβλήματα και πώς θα ε, παρεμποδίσουμε την επανάληψή τους. Γι' αυτό λοιπόν θα επανεξετάσουμε το σύμφωνο σταθερότητα για να εμβαθύνουμε την οικονομική επιτήρηση και να επεκτείνουμε εκτός του θέματος που αφορά στα ελλείμματα. Έχουμε ανάγκη από μηχανισμού για την επίλυση των κρίσεων. Εν συντομία θα πρέπει να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη βρίσκεται σύμπτωση των περιστάσεων και των κρίσεων και να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη Λισαβόνας. Γι' αυτό λοιπόν μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες της Κομισιόν και θα είναι τον επόμενο μήνα να υποβάλει μια έκθεση, μια ανακοίνωση μάλλον για την ενίσχυση των οικονομικών πολιτικών. Ε, γνωρίζουμε λοιπόν ποιο είναι το, το οικονομικό συμφέρον της Ευρώπης. Η Ευρώπη θα πρέπει να ενισχύσει το σύστημά της για να λάβει υπόψη όλες τις πιθανότητες κινδύνου και των οικονομικών ανισοτήτων και ανισορροπιών. Πρέπει να ενισχύσουμε τους ιστορικού μηχανισμούς αποκτώντας δομές πιο σταθερές και με έναν καλύτερο συντονισμό μπορούμε λοιπόν να επανέλθουμε σε ένα βιώσιμο δρόμο και να δημιουργήσουμε μια βάση για βιώσιμη ανάπτυξη. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, τους 18 τελευταίου μήνε κάναμε σημαντικέ πρόοδου στην υλοποίηση ενό χρηματοοικονομικού συστήματο πιο σταθερού και πιο υπεύθυνου. Πρέπει να ακολουθήσουν, να συνεχίσουμε αυτόν τον δρόμο, να καλύψουμε τι ελλείψεις που υπάρχουν στο επίπεδο κανονιστικό και να βεβαιωθούμε ότι θα μπορούμε να εποπτεύουμε αυτού του τομέα ο οποίο βρίσκεται σε εξελίξη. Τα εναλλακτικά λοιπόν κεφάλαια και τα επενδυτικά κεφάλαια ε, είναι κάτι στο οποίο η Κομισιόν πιστεύει πως ε, θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε έτσι ώστε μια νέα αρχιτεκτονική επιτήρηση και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού κλάδου θα θεθεί σε εφαρμογή το προσεχέ έτο. Το 2010 η Κομισιόν προτίθεται να παρουσιάσει πολλέ προτάσει ε, του λεγόμενου τομεί κλειδιά όπω τα παράγωγα ε, το ζήτημα εγγύησης ε, των ε, καταθέσεων και η προστασία από τις καταχρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να πρόσουμε ιδιαίτερη σημασία στην εποπτεία της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Θα πρέπει να εξετάσουμε επίσης και το θέμα των CDS και διάφορες άλλες συναλλαγές. Θα προβάλλουμε προτάσεις για το θέμα της πτώχευσης των τραπεζών. Κύριε Πρόεδρε κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε αμέσως με το να παρουσιάσουμε τη στρατηγική του 2020 αμέσως μόλις αναλάβαμε καθήκοντα. Πρέπει να ξαναφέρουμε την Ευρώπη στο σωστό δρόμο, στο δρόμο της έξυπνης βιώσιμης ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή. Πρέπει λοιπόν Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Κομισιόν, κράτη-μέλη να δημιουργήσουμε, να διατηρήσουμε αυτή την ορμή. Το να επιτύχουμε μια τέτοια κοινωνική οικονομία της αγοράς μέχρι το 2020 απαιτεί σοβαρές προσπάθειες από όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να έχουμε πραγματική προστιθέμενη αξία. Αυτός είναι ο στόχος των πρωτοβουλειών μας της ψηφιακής ατζέντας για την Ευρώπη, μιας πλήρους βιομηχανικής πολιτικής, ενός ευρωπαϊκού σχεδίου έρευνα και ανάπτυξη, μιας Ευρώπης που θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά του πόρου, νέε δεξιότητες, νεολαία εγκινήσει και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Εκεί μπορεί να κάνει τη διαφορά η Ευρώπη. Για να περάσουμε σε μια οικονομία που θα αντέχει στην κλιματική αλλαγή. Η καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής παραμένει πρώτη προτεραιότητα εσωτερικά και παγκοσμίας. Ο... Οι τομείς ενέργειας και των μεταφορών θα τύχουν ιδιαίτερης προσοχής καθώς και οι δύο παίζουν κρίσιμο ρόλο για να γίνουν ένα συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Η ενιαία αγορά ως αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών που θα προσφέρει δουλειές και ε, υπηρεσίες αγαθά σε ε, λογικές τιμές παραμένει βεβαίως ε, η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και βεβαίως η καινοτομία θα δημιουργήσει νέες δουλειές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να έρθει λοιπόν η ενιαία αγορά στον 21ο αιώνα αποτελεί προτεραιότητα της Κομισιόν η οποία θα καταθέσει νέες προτάσεις μέχρι το 2012. Αυτό είναι αντικείμενο έκθεσης ε, την οποία ζήτησα να προετοιμάσει ο Μάριο Μόντι και θα σας παρουσιάσουμε σύντομα. Δεν θα... Δεν χρειάζεται νομίζω να τονίσω ιδιαίτερα την σημασία της κοινωνικής ένταξης. Η Ένωση πρέπει να κοιτάξει ιδιαίτερα τους αδύναμους πολίτες της, να εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε ευκαιρία κοινωνικής συνοχής, να εκμεταλλευτούμε τους νέους τομείς που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Σημαίνει να δώσουμε στους ανθρώπους κατάλληλες δεξιότητες για να έχουμε υψηλά επίπεδα απασχόλησης και να διευκολύνουμε την οικονομική μετάβαση, να ξεπεράσουμε τον αντίκτυπο της κρίσης τους νέους για να μπορέσουν να περάσουν από την εκπαίδευση στην εργασία. Οπότε θα δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα καταπολέμησης της φτώχειας στο τρέχον ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης φτώχειας. Όλα αυτά βεβαίως συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των αρχών μας μιας οικονομικής και κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, όλα αυτά παραμένουν στο κέντρο της δράσης Κομισιόν. Η εφαρμογή του σχεδίου της Στοκχόλμης που θα υιοθετήσει η Κομισιόν αργότερα εντός της ημέρας σκοπεύει να διασφαλίσει πως τα Οφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης να είναι απτά από τους πολίτες. Οπότε θα πρέπει να εργαστεί η Κομισιόν προς αυτό. Βάζει τους πολίτες στο κέντρο των πολιτικών μας με το να διευκολύνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη και στο άνοιγμα μιας ασφαλούς Ευρώπης με ιδιαίτερο βάρος στην καταπολέμηση του διασυναριακού εγκλήματος και στην κοινωνική πολιτική μετανάστευση όσον αφορά τη δικαιοσύνη και τα εσωτερικά τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε περάσει από την εφαρμογή της ελεύθερης διακίνησης προσώπων σε μια κοινή πολιτική. Τα επιτεύγματα είναι εντυπωσιακά, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερο τώρα που βγαίνουμε από την κρίση να προωθήσουμε και να υπερασπιστούμε τις ευρωπαϊκές αξίες και να εκδιπλώσουμε όλο το δυναμικό που δημιουργεί η Συνθήκη της Λισαβόνας. Το σχέδιο δράσης περιέχει ένα κατάλογο μέτρων για να εφαρμόσουμε τις προτεραιότητές μας σε αυτόν τον τομέα, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η θέση ενισχύ της Συνθήκης Λισαβόνας μας δίνει τα εργαλεία για να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Ο αυξημένος ρόλος του Κοινοβουλίου η πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο. Σημαίνει πως θα έχουμε και καλύτερη συνοχή όσον αφορά τις αποφάσεις στο Συμβούλιο και βεβαίως ο έλεγχος από το δικαστήριο σημαίνει πως θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και ανησυχίες των πολιτών μας. Όταν κοιτάμε προς το 2020 πρέπει επίσης να δούμε κάποιες μακροχρόνιες τάσεις που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των πολιτών. Αν δράσουμε τώρα θα έχουμε τα ωφέλη στο μέλλον. Παραδείγματο χάρη θα ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση για το μέλλον των συντάξεων και θα αναλύσουμε επιλογές για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των συστημάτων συντάξεων. Βεβαίω, σε πολλού τομεί ε, πολλά από τα εργαλεία είναι εθνικά. Αυτό όμω δεν θα πρέπει να μα εμποδίσει να διασφαλίσουμε πώς θα συνεισφέρει στο μάξιμουμ η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των εξωτερικών. Ο νέος ρόλος της αντιπροέδρου της ε, Κομισιόν, της ΥΠΑ, της εκπροσώπου και η νέα υπηρεσία εξωτερικής δράσης σημαίνει πως θα έχουμε πιο ισχυρή εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Θα προωθήσουμε τις εμπορικές μας δράστερεότητες σε ζητήματα που αφορούν ε, από τις ε, ανισορροπίες μέχρι τις εμπορικές σχέσεις. Γενικότερα επίσης η Κομισιόν θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της γεωπολιτικής, της ενέργειας για να έχουμε ασφαλή βιώσιμη και φτηνή ενέργεια. Ένας άλλος στόχος της Κομισιόν είναι να διασφαλίσουμε την διεθνή ατζέντα της ανάπτυξης για να προετοιμάσουμε την σύνοδο των αναπτυξιακών στόχων του 2015 για να έχουμε μια κοινή θέση της Ένωσης εν ώψη της ε, συνάντησης ε, τον Σεπτέμβριο για, του ΟΗΕ για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας για να έχουμε νέους τέτοιους στόχους το 2015. Και έτσι δείχνουμε συγκεκριμένα την αλληλεγγύη μας με τους πιο ευάλωτους σε αυτόν τον κόσμο. Τέλος, θα υιοθετήσουμε μέχρι το τρίτο τρίμηνο μέχρι το τρίτο τρίμηνο αυτού του έτους νέους στόχους για τον προϋπολογισμό. Παράλληλα θα αξιολογήσουμε το κλειδιά όπως η Γεωργία και άλλοι τομείς σας διαβεβαιώνω λοιπόν πως ε, θα σας εμπλέξει η Κομισιόν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πριν τελειώσω, θα ήθελα να εξηγήσω κάποιες καινοτομίε στο πρόγραμμα της Κομισιόν. Το πρόγραμμα αυτό και τα μελλοντικά προγράμματα πρέπει να αποτελούν ένα ευρύ πλαίσιο για να μπορέσουν να βασιστούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οπότε πρέπει να είμαστε πιο πολιτικοί και να αντικατοπτρίζεται εδώ πέρα η πρόκληση και η κλίμακα των πρωτοβουλειών μας. Πρέπει λοιπόν τα μελλοντικά μας προγράμματα να επιδεικνύουν συγκεκριμένα την ειδική εταιρική σχέση που θέλουμε να έχουμε εγώ και όλοι οι Κομισιόν με το Κοινοβουλίο σας. Το πρόγραμμα αυτό έχει 34 στρατηγικές πρωτοβουλίες που δεσμευόμαστε να καταθέσουμε πριν από το τέλος Σεπτεμβρίου. Θα συμφωνείτε πως είναι φιλόδοξο πρόγραμμα για 8 μήνες. Ταυτόχρονα συμπεριλαμβάνει και άλλες πρωτοβουλίες για το 2010 και μετά. Ο ενδεικτικός αυτός κατάλογος συμπεριλαμβάνει πρωτοβουλίες που σκοπεύει να δει η Κομισιόν τα ερχόμενα χρόνια. Δεν σημαίνει πως ε, θα οδηγηθούμε σε συγκεκριμένες προτάσεις καθώς πρέπει να ακολουθήσουμε και τις αρχές της καλύτερης ρύθμισης και να δούμε σε ποια θέματα πρέπει να προχωρήσουμε και σε ποια όχι το πρόγραμμα αυτό θα αναθεωρείται κάθε χρόνο για να βρούμε νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες και να προσαρμοζόμαστε. Η συνεχής αυτή προσέγγιση σημαίνει πως θα έχουμε διαφάνεια και προβλεψιμότητα και την απαραίτητη ευελιξία για να μπορούμε να αντιδρούμε στις εξελίξεις. Καθώς, όπως μάθαμε τελευταία χρόνια, πρέπει να προβλέπουμε το απρόβλεπτο. Αυτό σημαίνει πως στρατηγική μας στόχη δεν μπορεί πλέον να είναι θέσφατα. Πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται. Οπότε είναι ένα απαραίτητο αλλά και φιλοδοξό πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια. Ρεαλιστικό, εάν είναι βεβαίως όλα τα θεσμικά οργανά πρόκειται να συνεργαστούν για να έχουμε αποτελέσματα για τους πολίτες. Και βεβαίως ε, δεν γίνεται να συνεχίσουμε όπως συνεχίζαμε, αν είναι να έχουμε μια αλλαγή το 2010 και βεβαίως φιλόδοξο γιατί πρέπει να έχουμε περισσότερη Ευρώπη για να έχουμε αποτελέσματα για τους πολίτες. Αυτό αναμένουν από εμάς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε για την ε, διεξοδική παρουσίαση των σημαντικότερων πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο οκτάμινο. Τώρα θα ακούσουμε τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Πάντως, η στρατηγική εταιρική σχέση που αναφέρατε, κύριε Πρόεδρε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντική. Γιατί γίνεται ένας διαχωρισμός μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, αλλά η συνεργασία μας ε, έχει νευραλική σημασία και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό ε, συμφωνούμε με την ε, επισήμασή σας για την αναγκαιότητα στενών επαφών μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και η αθρώα προσέλευση επιτρόπων σήμερα στην Ολομέλεια είναι περίτρανη απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εννοεί αυτή την ανάγκη για στενή συνεργασία. Θα ακούσουμε τώρα εκ μέρου ε, των πολιτικών ομάδων του εκπροσώπου ε, τον αντιπρόεδρο πρώτα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, τον κύριο Γιώζεφ Σάγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζουμε το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν και χαιρόμαστε για το ότι ε, προγραμματίζεται συνεργασία με το Κοινοβούλιο και για το ότι είστε εδώ. Αλλά είναι κρίμα το ότι χάσαμε ήδη κάποιους μήνες. Φέτος η συνθήκη της Λισαβόνας έτεθην ισχύει καθυστερημένα και αυτό σημαίνει πως δεν είχαμε ισορροπία μεταξύ της ε, υλοποίησης ε, και του σχεδιασμού του νομοθετικού προγράμματος και ελπίζουμε να αποκατασταθεί η συνθήκη της Λισαβόνας, τέθη ενισχύ, δεν έχουμε καμία αντίρρηση ούτε το Κοινοβούλιο, ούτε το Συμβούλιο, ούτε η Κομισιόν και δεν έχουμε λόγο να μην ξεκινήσουμε αμέσως τη δουλειά. Πρέπει να ξεκινήσουμε να εκφράζουμε τα συμφέροντα των πολιτών να φροντίζουμε για την δική τους ε, την ευημερία. Βεβαίως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει συντάξει δύο καταλόγους όσον αφορά το πρόγραμμα και εδώ πέρα βέβαια έχουμε αναφέρει και τις δραστηριότητες που αναμένουμε από σας. Θέλουμε από την Κομισιόν να χρησιμοποιήσει έναν άλλο, μια άλλη προσέγγιση. Δεν θέλουμε να κάνετε τις, να έχετε υλοποιήσει μόνο το 40% των νομοθετικών σας προτάσεων μέχρι τον Οκτώβρη, γιατί αν ε, μείνουν έτσι τα πράγματα δεν μπορεί και το Κοινοβούλιο να εκφραστεί για αυτές τις προτάσεις σας και θα θέλαμε να μην κάνετε όπως έκαναν τα κομμουνιστικά κράτη με τα πενταετή προγράμματα γιατί εκεί πέρα βεβαίως στο τέλος εφαρμόζονταν μόνο ένα κλάσμα αυτών των προγραμμάτων. Πολλές κυβερνήσεις τώρα ε, βρίσκονται σε κρίση γιατί έλεγαν ψέματα για τα ελλείμματά τους, έκρυβαν τα στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει όλοι στην ίδια βάρκα είμαστε. Ουγγαρία, Ελλάδα ε, πέρασαν μια παρόμοια κρίση σε μια δύσκολη κατάσταση ε, βρέθηκαν και θέλουμε από την Κομισιό να κατονομάσει τις χώρες που δεν τηρούν τις κανόνες ο Κόμις Σέσελη είχε πει πως όσοι κρύβουν την αλήθεια κάνουν χειρότερο κακό. Μη με παρεξηγήσετε. Δεν θέλω εγώ, δεν θεωρώ την Κομισιόν υπεύθυνη. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών είναι υπεύθυνε. Αλλά η Κομισιόν έπρεπε να έχει δει τα σημάδια. Οπότε, τι πρέπει να κάνει η Κομισιόν. Θέλουμε από την Κομισιόν να επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα για την αποκατάσταση της οικονομίας, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό πρέπει να αποτελεί την κατευθυντήρια γραμμή μας. Εάν είναι να μιλήσουμε στους πολίτες, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια γλώσσα που την καταλαβαίνουν οι πολίτες. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα πρώην κομμουνιστική. Οπότε δεν μπορώ εγώ να μιλάω για πενταετή προγράμματα. Για πενταετή πλάνα. Μπορούμε τη στρατηγική 2020 να την πούμε στρατηγική για τις ε, θέσεις εργασίας, στρατηγική της Στοκχόλμης, να την πούμε για την ασφάλεια των πολιτών, να διαλέγουμε προσεκτικά τις λέξεις. Επίσης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκεί πέρα πρέπει να δημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας και δεν θέλουμε το πρόγραμμα αυτό για τη δημιουργία θέσεων εργασίας να υιοθετηθεί χωρίς ε, κριτική από πλευράς του Κοινοβουλίου. Όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να φροντίσουν για περισσότερες θέσεις εργασίας και να μάθουμε από τα λάθη της στρατηγικής της Λισαβόνας. Επίσης, ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Έχουμε και κοινέ αξίες. Πρέπει να τηρήσετε τις αξίες μας. Την κοινή ευρωπαϊκή ιστορία, την προστασία των μειονοτήτων. Εμείς θα σας υποστηρίξουμε, αλλά θα ασκήσουμε και κριτική. Please. Σας ευχαριστώ για την ομιλία σας, αλλά παρακαλώ μην παραβαίνετε το χρόνο που έχει ο καθένας στη διάθεσή του. Το λόγο κύριος Χάνες Βόποντα, ο αντιπρόεδρος ε, της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες ε, και κύριοι Επίτροποι. Σας ευχαριστώ που ήρθατε τόσο πολύ, κάτι το οποίο δεν μπορώ να πω για τους συναδέλφου μου. Και δεν είναι όλοι οι απόντες απόντες θα έπρεπε να είναι εδώ. Δεν είναι γιατί δεν μπορούν να έρθουν. Δεύτερον, βεβαίω ε, υπάρχουν και οι λεπτομέρειες που θα δείτε στο κοινό μας ψήφισμα. Τώρα, πού συμφωνούμε. Πράγματι πρέπει να δούμε την ανταγωνιστικότητα, την αηφορία, την κοινωνική δικαιοσύνη. Και βεβαίως εδώ πέρα βλέπετε πως έχουμε μια ανεργία η οποία αυξάνεται και είπατε πως πρέπει να καταπολεμήσουμε και την φτώχεια, κάτι το οποίο δεν ξέρω εάν το κάνουν όλοι οι αρχηγοί κυβερνήσεων. Πώς να γίνουν όμως όλα αυτά όταν μειώνονται οι προϋπολογισμοί. Βεβαίως πρέπει να γίνει αυτό, αλλά πρέπει να λάβει και η Κομισιόν υπόψη ότι αυτό πρέπει να γίνει με μια χρονική ακολουθία η οποία δεν θα, θυσιάσει τους άλλους μας στόχους, δηλαδή την καταπολέμηση της φτώχειας. Και επειδή είχαμε και την σύνοδο της Κόρδομπας, στην οποία δεν ήσταν εσείς βεβαίως, αλλά, αλλά μέλη της ε, Κομισιόν, Αντιπρόεδρο νομίζω και ο επίτροπο για τα Κοινωνικά. Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Είχα πάει πρόσφατα και είδα στη Σερβία το πώς ζουν οι Ρώμα. Πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα ε, για τη σημερινή Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την καταπολέμηση της στόχης και των διακρίσεων στην Ευρώπη. Μια που μιλήσαμε λοιπόν για τον περιορισμό των προϋπολογισμών, να πούμε πώς χρειαζόμαστε το αντίθετο. Χρειαζόμαστε επενδύσεις. Το συζητήσαμε με τον κύριο Κάλλας. Δεν υπάρχουν επενδύσεις π.χ. στα διευρωπαϊκά δικτύα και βλέπουμε σήμερα τι προβλήματα έχουμε. και βλέπετε πώ δεν είχε ακολουθεί. Ε, βλέπετε παραδείγματο χάρη τι είχε γίνει όταν είχε προταθεί το σχέδιο Delors. Πρέπει λοιπόν να τα δείτε αυτό και στο τωρινό και στα επόμενα σχέδια του προπολογισμού. Χρειαζόμαστε αυτή την εταιρική σχέση γιατί βλέπετε πώ θέλει να περικόψει το Συμβούλιο του προπολογισμού. Κύριε Πρόεδρε, επίση μιλήσατε για την έκθεση Μόντι. Πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντική και σημαντικό το να θέσετε τον κύριο Μόντι, ο οποίο είναι ειδικό, αλλά Εάν μιλάμε για ενιαία αγορά, για την οποία μιλήσατε, πρέπει να μιλήσουμε και για την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Εδώ πέρα λοιπόν παίζουν ρόλο οι δημόσιες υπηρεσίες. Είπατε πώς θα έρθετε με μια οδηγία πλαίσιο. Δεν θέλουμε τώρα να δούμε όλες τις λεπτομέρειες εδώ πέρα, αλλά πρέπει ακριβώς στις κοινοφελείς υπηρεσίες να υπάρχει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα. Και εδώ πέρα είναι το πρόβλημα το οποίο έχουμε πάλι. Τι γίνεται, όπως παραδείγματο χάρη, με τους σιδηρόδρομους. Είτε είναι ιδιωτικές είτε κρατικές εταιρείε. Αλλά πρέπει βεβαίως να υπάρχει διασφάλιση και ρύθμιση με μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Και έρχομαι στο τελευταίο και αποφασιστικό νομίζω ζήτημα. Μιλήσατε για την οικονομική κρίση Μιλήσαμε για την Ελλάδα και άλλες χώρες που βρίσκονται σε κρίση. Την τελευταία φορά διαπιστώσαμε στη συζήτηση με τον κύριο Φαν Ρόμποϊ πως ε, αυτά τα οποία έκανε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ήταν και πολύ ικανοποιητικά. Εάν τα είχαμε κάνει πριν από δύο ή τρεις μήνες θα μπορούσε να είχε αποφύγει τα υψηλά επιτόκια η Ελλάδα. Το είπατε, το το υπονοήσατε. Αλλά χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Χρειαζόμαστε την ισχυρή φωνή της Κομισιόν. Είναι θέμα δικαιοσύνης. Το θέμα δεν είναι γιατί υπάρχουν παρεξηγήσεις εδώ πέρα όταν, φτάσουν η, όταν φτάσει η κρίση να επέμβουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να την προλάβουμε μέσω της επιτήρησης των χρηματαγορών, των εξελίξεων στου ε, προπολογισμού. Όχι, όχι λένε οι κυβερνήσεις, δεν μπορείτε να δείτε τα στατιστικά μα στοιχεία. Δεν είναι αποδεκτό αυτό. Εάν θέλουμε να εμποδίσουμε αυτά τα οποία συνέβησαν τους τελευταίους μήνες και έτος, πρέπει να το δούμε. Γιατί να κρύψει τα στατιστικά, τη στοιχεία και τον προπολογισμό τη μια κυβέρνηση. Βεβαίω έχει κάποιο χώρο ελιγμών, αλλά ειδικά εντός της Ευρωζώνης πρέπει να υπάρχει νομίζω και μια συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς στόχους. Τώρα φτάνουμε στην ειδική σχέση που αναφέρατε. Είμαστε διατεθειμένοι, αλλά αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή θέση και του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Διαπραγματευόμαστε αυτές τις μέρες για τη Συμφωνία Πλαίσιο. Καθορίζει κάποιες λεπτομέρειες, αλλά το πνεύμα της Συμφωνίας ποιο είναι. Το πνεύμα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Είναι πως όταν θέλουν κάποιοι κυβερνήσει να εκμεταλλευτούν τις συνθήκες της Λισαβόνας για να ενισχύσουν τη δική τους θέση. Όχι. Πρέπει να ενισχυθεί η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Εμείς οι δύο πρέπει να αγωνιστούμε για την ισχυρή Ευρώπη έναντι κάποιων αρχηγών κυβερνήσεων. Και είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε για την ομιλία σας και σας ευχαριστούμε θερμά γιατί σεβαστήκατε ευλαβικά το χρόνο σας και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη διεξαγωγή της συζήτησης. Η κυρία Μαρία Ντεσαρνέ. από τους φιλελεύθερους και δημοκράτες. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρά είναι άτολμο το πρόγραμμα το νομοθετικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεδομένων των προκλήσεων. Περιμένουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολλά δε μάλλον που αυτό είχατε εξαγγείλει αρχικά. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοπιστωτική ρυθμίση, αντιλαμβάνομαι τα μέτρα του κύριου Μπαρνιέ, βαίνουν προ τη σωστή άγουσα, αλλά και αυτά θα μπορούσαν να είναι πιο παράτολμα και φιλόδοξα. Για παράδειγμα, διαχωρισμό των τραπεζικών δραστηριοτήτων, ε, τη φορολογία των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή μεγαλύτερη ρύθμιση για τα παράγωγα όπως ε, σκέφτονται οι ΗΠΑ. Ακόμη πιο σημαντικό για μένα όμω είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να δώσουμε έμφαση και προνόμια στην πραγματική οικονομία και στις ε, βιώσιμες επενδύσεις που αυτές είναι που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε πολύ συγκεκριμένα σχέδια προς αυτή την κατεύθυνση, κάτι που δεν βλέπω στο νομοθετικό πρόγραμμα. Χρειαζόμαστε φυσικά και μεγαλεπίβολα σχέδια. Και Νομίζω ότι σήμερα είναι κατάλληλη στιγμή για να ξαναδώσουμε όθηση στα προγράμματα της ε, υπέρ των σιδηροδρόμων, γιατί 28.000 ε, πτήσεις ε, κάθε μέρα ακυρώνονται. Νομίζω ότι επιτέλους πρέπει να δώσουμε έμφαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Χρειαζόμαστε όμως και καλύτερο χρηματοοικονομικό και δημοσιονομικό συντονισμό και μια πραγματικά δημοσιονομική διακυβέρνηση και χρηματοπιστωτική. Ελπίζω να το λάβει από αυτό υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, χρειαζόμαστε δημοσιονομικό συντονισμό, οικονομικό συντονισμό και βιομηχανικό συντονισμό. Θα πρέπει να ιδρύσουμε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και να το εφοδιάσουμε με μέτρα εξυγίανση ε, των ε, εθνικών δημοσιονομικών ε, καταστάσεων. Επίση χρειαζόμαστε και μια φορολογική σύγκληση, για παράδειγμα εταιρικό φόρο, φόρο τη επιχειρήση. Θα πρέπει επίση να επεξεργαστούμε καλύτερα τον ε, κοινοτικό προπολογισμό. Νομίζω ότι έτσι θα μπορούσαμε να ξαναβρούμε το δρόμο τη ανάκαμψη. Σε ό,τι αφορά τη μελλοντική στρατηγική για το 2020, σα θέρμο παρακαλώ μην καταλήψετε κάποιου ποσοτικοποιημένου στόχου ε, για τη φτώχεια και την παιδεία. Νομίζω ότι έτσι θα τυχείτε τη αμέρη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί αυτό χρειαζόμαστε, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Αυτό μα είναι προσφυλέ. Σα ευχαριστούμε κύριε Τεσσαρνές. Το λόγο έχει η κυρία Ρεμπέκα Χάρμς, που είναι συμπρόεδρος των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι Επιτροπή. Θα ήθελα βεβαίω, ε, το σεβασμό τον οποίο επιδεικνύεται να τον ανταποδώσει και το Κοινοβούλιο με περισσότερες ε, παρουσίες. Τώρα το πρόγραμμά σας βεβαίω είναι ευρύτατο και περιέχει τίτλους που ακούγονται πολύ φιλόδοξοι. Π.χ. ήδη στην εισαγωγή μιλάτε για μία νέα εποχή. Δεν ξέρω εάν ε, μετά οι λεπτομέρειες κάτω από αυτούς τους μεγάλους τίτλους ανταποκρίνονται σε αυτές τις ε, απαιτήσει. Εξακολουθεί να υπάρχει κλιματική κρίση, χρηματοπιστωτική κρίση. Η Ελλάδα έδειξε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν έχει μόνο μια μεγάλη οικονομική ψαλίδα αλλά και ένα κοινωνικό χάσμα. Οι συνθήκες μεταξύ Βορρά, Νότου ή Ανατολής Δύσης είναι διαφορετικές ειδικά όσον αφορά τον τομέα κοινωνικής Ευρώπης και περισσότερης δικαιοσύνης μπορώ να συμφωνήσω με τον κύριο Σβόμποντα. Πρέπει να εργαστούμε ήδη αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας και ε, έχουμε ως εργαλεία φτάνουν για να καταπολεμήσουμε ε, την ε, φτώχεια. Τώρα αν το κάνουμε δεν είμαι τόσο πεπισμένη. Τώρα για την κρίση, για την οικονομική ολοκλήρωση. Αυτό το οποίο βρίσκουμε σωστό για την οικονομική ολοκλήρωση είναι πως γίνονται νέες προτάσεις για την φορολόγηση των επιχειρήσεων. Εμείς είμαστε υπέρ, ήμασταν ανέκαθεν υπέρ, είμαστε επίσης υπέρ της φορολόγησης της ενέργειας. Βασιστείτε πάνω μας εάν κάνετε κάτι τέτοιο αλλά δεδομένων των εμπειριών που είχαμε με την ε, χρηματοπιστωτική κρίση, αυτό το οποίο δεν υπάρχει είναι ένας ξεκάθαρος στόχος για ένα φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Εντάξει, μπορούμε να τα αφήσουμε στα καρατιμέλη, αλλά εδώ πέρα ισχύει αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σάιερ. Καμιά φορά πρέπει να έχετε πιο συγκεκριμένες απαιτήσει και να παλέψετε για αυτές. Το ότι δεν αντιδράσαμε παρκώς στην περίπτωση της Ελλάδας είναι σαφές. Δεν έγινε καμία πρόταση για ευρώ ομόλογα απαράδεκτο. Κύριε Μπαρόζο, μιλήσατε επίσης και κάνατε μια καμπάνια για τις κοινοφελείς υπηρεσίες. Πράγματι, και εδώ πέρα νομίζω πως ε, κάτω από τον τίτλο που λέτε ότι ο άνθρωπος είναι στον κέντρο, οι υπηρεσίες αυτές κοινή ωφέλειας και ε, η ρύθμιση που θέλουμε να επιτύχουμε πράγματι δεν υπάρχει και εδώ πέρα εάν δεν το κάνετε θα παραβιάσετε την προσωπική σας υπόσχεση. Όσον αφορά δε την προστασία του κλίματος. Οι διαφορετικές γενικές διευθύνσεις που ασχολούνται με αυτό επεξεργάζονται σενάρια με διαφορετικούς στόχους για το 2050. Μιλάμε στην συγκοινωνίες για μείωση κατά 70%, ενέργειες 75%. Εντάξει, ε, είναι φιλόδοξη, αλλά σε καμία γενική διεύθυνση δεν παίζει κανένα ε, ρόλο το μπαλί, ο στόχος των δύο βαθμών Κελσίου. Τιος είναι ο στόχος της ευρωπαϊκής κλιματικής διπλωματίας εάν δεν προωθούμε τον παλί ή τις αποφάσεις των G8. Αυτά τα οποία είναι στο πρόγραμμα λοιπόν δεν ε, επαρκούν για να είμαστε επιτυχημένοι στη Βόνη, στον Κανκούν ή στην Νότια Αφρική. Δεν επαρκούν. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Το λόγο κύριο Τίμωθη Κίρκοπφ, ο πρόεδρο ε, των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σα υπενθυμίσω τα διδάγματα του προγράμματο του 1992. Για να υλοποιήσει στόχου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να θέσει μία προτεραιότητα και να επικεντρωθεί σε μία πολιτική κάθε φορά η απόπειρα ίδρυση εσωτερική αγορά ήταν μεγαλεπίβολο στόχο, εύκολα αντιληπτό, ε, που τον κατανοούσαν και οι Ευρωπαίοι πολίτε. Έκτοτε όμω και πολύ συχνά βλέπουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συσσωρεύει τη μία πρωτοβουλία μετά την άλλη, χωρί όμω ε, να φέρνει αυτά αποτελέσματα, ελπίζοντα μόνο να γίνει δημοφιλή. Ήταν ε, λάθο αυτή η προσέγγιση. Χαίρομαι για την ακατεύθυνση που φαίνεται ότι ακολουθεί ο πρόεδρο Μπαρόζο. Η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε βαθύτατη κρίση και μόνο συγκεκριμένε δράσει και συνεπεί θα αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Δεν μιλάω μόνο για την κρίση εξαιτία τη αποτυχία του τραπεζικού συστήματο ή την απρόσμενη κρίση που είχαμε στι ενέργειε μεταφορέ. Έχουμε και μια λανθάνουσα κρίση τη ευρωπαϊκή οικονομία που μένει πίσω όσο αφορά την ανταγωνιστικότητά τη απέναντι στι ισχυρότερε οικονομίε τη Ασία, για παράδειγμα, ή των ΗΠΑ θα πρέπει να προσθέσουμε κάποιες λεπτομέρειε στη στρατηγική του 2020. Πάντως η γενική κατεύθυνση της στρατηγικής του 2020 είναι σωστή. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική για ευφυή, βιώσιμο και συμμετοχικό, συμμετοχική πρόοδο και ανάπτυξη. Αξία όλοι αυτοί οι στόχοι και έτσι θα πρέπει από αυτά θα πρέπει να καθοδηγεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φυσικά όλα αυτά εξαρτώνται από τι επιτυχημένε επιχειρήσει και του επιχειρηματίε. Αυτοί είναι που δημιουργούν πλούτο και θέσει απασχόληση. Αυτή είναι η καλύτερη πολιτική καταπολέμηση τη ένδυα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι σύμμαχος αυτών των επιχειρήσεων και όχι ε, αντίπαλός τη. Θέλουμε να επεκτείνουμε την εσωτερική ναι. αγορά με φύση, διατάξει, να εξασφαλιστεί τη εφαρμογή των κανόνων με θεμητό και δίκαιο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ελαφρυνθεί η γραφειοκρατία και το περιττό διοικητικό άχθο, Θα πρέπει να ξεχρονίσουμε την αγορά εργασία, να δώσουμε έμφαση στην κατάρτιση και να καταργήσουμε τους εμπορικούς φραγμούς. Θέλουμε μια δυναμική ευρωπαϊκή οικονομία και αν αυτό ε, επιδιώξει ο κύριος Μπαρόζο θα Τύχη τη αμέριστη υποστήριξή μα. Φυσικά δεν θα πρέπει να αμελούμε τι ευθύνε των κρατών μελών. Έχουμε την πρόταση για την Ευρώπη των πολιτών. Κάποια ε, στοιχεία του προγράμματο Στοκχόλμη. επίση τι κοινέ ε, αγορέ ε, γεωργία και πολιτική. Θέλουμε όμω πολύ πιο δίκαιε λύσει για του γεωργού και του ελλεί μα. Δεν συμφωνούμε ότι οι κοινέ ε, πρωτοβουλίε γίνονται από τα κράτη-μέλη που γίνονται από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλυθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να καταληφθούν από τα κράτη-μέλη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η ως λύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και η επικουρικότητα. Θέλουμε αυτά αποτελέσματα και ελπίζουμε ότι η νέα Επιτροπή του κυρίου Μπαρόζο ε, να δράξει την ευκαιρία του νομοθετικού αυτού προγράμματος και να εξασφαλίσει μια ισχυρή παρουσία της Ευρώπης, ε, να εξασφαλίσει την οικονομική ανάκαμψη και μια βιώσιμη ευημερία και αηφόρα ευημερία στους χαλεπούς καιρούς που βρίσκονται μπροστά μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ομιλία σας. Τώρα εκ μέρους ε, της ΓΚΟΕ το λόγο έχει ο κύριος Μιγγέλ Πόρτας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο τίτλος του νομοθετικού προγράμματος που εξετάζουμε σήμερα είναι είναι και η ώρα της δράσης. Χρειάστηκαν όμως πέντε μέρες για να διοργανωθεί μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ των υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ωραία τα λόγια, αλλά χρειαζόμαστε έργα. Είναι και η ώρα της δράσης. Τι σημαίνει αυτό, ότι μέχρι τώρα είμαστε αδρανείς. Ο τίτλος αυτός μήπως είναι μια αυτοκριτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή μήπως αυτός ο τίτλος όπως και όλοι οι άλλοι τίτλοι των γραφειοκρατικών ανακοινώσεων είναι ένα κενό γράμμα, ε, είναι μία δράνεια που κρύβεται πίσω από ένα σωρό λέξεων και αγαθών προθέσεων. Μιλήσαμε για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Μιλάτε για μία πρωτοβουλία για να εξασφαλιστεί καλή κατανομή των ε, ωφελών της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Μήπως και αυτό είναι πλάκα που μας κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι πρωτοβουλία είναι αυτή και πώς μπορεί να αντισταθμίσει την ε, απόσυρση των κοινωνικών ε, επιδοτήσεων που κάνουν τα κράτη-μέλη στο βωμό και με το πρόσχημα των προγραμμάτων σταθερότητας. Τι κατανομή ε, πλεονεκτημάτων θα γίνει αφού δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Πώς θέλετε να μειώσετε τον αριθμό των φτωχών αν δεν αγγίξετε τα κέρδη των πλούσιων και των πάπλουτων διαφωνούμε ως προς την πολιτική με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί ε, ε, επανέρχεται η δικτατορία του ελίματος που εγκλωβίζει τις οικονομίες, περικόπτει τους μισθούς, τα επιδόματα και τις δημόσιες ε, επενδύσεις σε κοινοφελείς υπηρεσίες. Αυτή είναι συνταγή για περισσότερη ανεργία και όχι περισσότερη απασχόληση. Είναι και, η ώρα της δράσης μας, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύει λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανασκουμποθεί και να συσπηρώσει τις δυνάμεις της για να αντιμετωπίσει την κρίση. Ρωτήστε τους Έλληνες αν είναι αυτή της γνώμης. Αν ήμασταν άμεση στη δράση μας και αν ήμασταν δίκαιοι. Πότε θα συστηθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. Ρωτήστε τους Πορτογάλους ε, που έχουν χρέη και πώ ακούν τους επιτρόπους που μιλούν για την οικονομία. Ρωτήστε τους Ευρωπαίους πολίτες γιατί η κατάσταση έχει όσα έχει. Γιατί μερικές φορές ακούγοντας τα λόγια μας χαμογελούν και κοροϊδεύουν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λέει ο κύριος Πρόεδρος. Το λόγο ο κύριος Φιωρέρο Προβέρα από την Ελευθερία και Δημοκρατία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, που αποτελούν το 99% του ε, παραγωγικού ιστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν ανάγκη από τέσσερα βασικά στοιχεία. Με πρόσβαση στις πιστώσεις, ε, μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας, λιγότερο γραφειοκρατία προκειμένου να ιδρυθούν και να τύχουν διαχείριση και τέλο προστασία από την του ανταγωνισμό. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τι εργασίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, βελτίωση της γραφειοκρατίας με την κατάρριξη 1.200 ε, ε, γραφειοκρατικών πράξεων που απαιτούνται. Ε, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι η κατάσταση σε επίπεδο διεθνού εμπορίου. Σε αυτή την περίοδο κρίση χρειάζεται το σύστημα εμπορική άμυνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να ενισχυθεί. Οι επιχειρήσει δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ που εφαρμόζουν ορισμένε αναδυόμενε οικονομίε όπω ε, αυτή τη Κίνα, όπου το κόστο εργασία είναι πολύ ιδιαίτερα χαμηλό, δεν υπάρχει κοινωνική προστασία αλλά και ούτε υψηλά πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα πρέπει να επένδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η καταπολέμηση των απομιμήσεων και των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν υπάρχει καμία πρωτοβουλία στο πρόγραμμα της Κομισιόν σχετικά με τα όσα προβλέπει η συνθήκη τη Λισαβόνα για την πολιτική συνοχή. Για πρώτη φορά το άρθρο 174 της συνθήκης αναγνωρίζει τον συγκεκριμένο ρόλο των ορεινών περιοχών που αποτελούν το 40% του εδάφους μας και κατοικούν άνω των 90 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Θα ζητώ λοιπόν να συμπεριλάβετε στο μελλοντικό ε, πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομοθετικό μια πρόταση πλαίσιο για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της προστασίας των ορεινών περιοχών και για να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που προσφέρουν οι ορεινοί όγκοι. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος ε, των μη εγγεγραμμένων το λόγο έχει ο κ. Μπρόντσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο πρόγραμμα εργασίας Κομισιόν για το 2010 λέει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει μακροπρόθεσμες ε, προκλήσεις όπως η παγκοσμιοποίηση και να ξαναβρει την ανταγωνιστικότητα. Δεν την αντιμετωπίζει, την έχει αγκαλιάσει. Επιτρέπει σε μια πλημμυρίδα εισαγωγών να καταστρέψουν το εμπόριο στην Ευρώπη. Η μόνη ανταγωνιστικότητα που μπορούμε να έχουμε είναι να μειώσουμε τους μισθούς στα επίπεδα αυτών των χωρών. Εγώ δεν είμαι καν υπέρ του να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να ήμουν υπέρ θα έλεγα πως οι διοικούντες έχουν προδώσει τους ανθρώπους. Δεν είναι μια οικονομική και Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά μια παγκόσμια ένωση που προσπαθεί εδώ πέρα να επιβάλλει τις εισαγωγές άλλων κρατών. Πρέπει τα κυρίαρχα κράτη να ξαναφτιάξουν την παραγωγική τους φάση όσον αφορά τους ευρώφιλους. Είτε ενωμένη είτε χωριστά η Ευρώπη δεν θα προστατεύσει την ε, παραγωγή της ε, και τη γεωργία της από τις εισαγωγές και αυτό είναι κίνδυνος για την ίδια. Είτε θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε είτε θα καταστραφούμε όλοι από την παγκοσμιοποίηση. Πρέπει επίσης να δούμε τους κινδύνους της δημογραφικής γύρανσης. Οπωσδήποτε είναι ανησυχία ή γυραιοί πληθυσμοί σε πολλές χώρες. Πρέπει όμως να δούμε γιατί εμφανίστηκαν αυτά τα προβλήματα καθώς πολλές γυναίκες ακολουθούν την καριέρα τους είναι δικαίωμά του βεβαίω να κάνουν αυτή την επιλογή, αλλά πάρα πολλέ άρε εργάζονται γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Εργάζονται για να πληρώσουν του λογαριασμού, όχι γιατί περιφρονούν τη μητρότητα. Οπωσδήποτε αυτό έχει αντίκτυπο στο ρυθμό γεννήσεων που έχει πιεστεί από τις οικονομικές δυνάμεις. Αυτό όμω δεν σημαίνει πως πρέπει να αφήνουμε τις οικονομικές δυνάμεις να κάνουν ό,τι θέλουν. Μπορεί να υπάρξει πίεση να αντιδράσουμε σε, αυτός και, σε αυτές και ανάλογα θα μεταβληθεί και η δημογραφική κατάσταση. Η ιδέα ότι μπορούμε να εισάγουμε μεγάλες οικογένειες από τον τρίτο κόσμο ως υποκατάστατο των, παιδιών που θα γεννιούνται στην Ευρώπη δεν είναι σωστή. Δεν είναι παλτά τα οι πολιτισμοί τα οποία θα τα φοράνε στο σημείο εισόδου και θα τα αποκτούν τον πολιτισμό αυτό με τα χαρτιά. Τα παιδιά λένε των μεταναστών αυτών είναι όσο Ευρωπαίοι όσο και οι αυτόχθονες πληθυσμοί. Όχι. Οι πολιτισμοί δημιουργούνται από του ανθρώπου και όχι αντιστρόφω. Δεν είμαστε προϊόν του πολιτισμού μα. Ο πολιτισμό είναι προϊόν των λαών μα. Το να αντικαθιστούμε του Ευρωπαίου με ανθρώπου από τον τρίτο κόσμο σημαίνει πω η Ευρώπη θα αντικατασταθεί από τον τρίτο κόσμο. Αργά αλλά σταθερά υπάρχει εθνοκάθαρση τη Ευρώπη και εξαφανίζονται οι Ευρωπαίοι. Σα ευχαριστώ. Το λόγο θα δώσω τώρα στον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να δευτερολογήσει. Κύριε Μπαρόζο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά δεν μιλάω για αυτούς που είναι πολέμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως γενικά εγώ διέκρινα μία σύγκληση και μία σύμπνοια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αν υπάρχει ένα κοινό στοιχείο που διέγνωσα στους εκπροσώπους των πολιτικών δυνάμεων είναι η ιδέα της φιλοδοξίας, ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία. Και από αυτή την άποψη θα καταγράψω ορισμένες ιδέες ε, που άκουσα και με τις οποίες συμφωνώ. Ο κύριος Σάγερ μίλησε για την ανάγκη να αποφύγουμε το μοντέλο των πενταετών προγραμμάτων των κομμουνιστικών καθεστώτων. Γι' αυτό ακριβώς εμείς θέλουμε να διαφυλάξουμε μία ελαστικότητα. Είναι σημαντική αυτή η ελαστικότητα και μας επιτρέπει να προσαρμοζόμαστε σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Φυσικά, θα πρέπει να διευκρινίσω απαντώντας και στον κύριο Σάγερα αλλά και στον κύριο Σφόμποντα ότι έχουν δίκιο που ζητούν ε, μεγαλύτερη δραστηριοποίηση σε θέματα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στηλίτευσαν την απροθυμία των κρατών μελών ε, σε ό,τι αφορά ένα ενισχυμένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιτήρηση των ε, εθνικών ε, λογαριασμών στην προηγούμενη επιτροπή είχα προτείνει ένα κανονισμό, συγκεκριμένο κανονισμό για να αυξηθούν τα, οι, οι αρμοδιότητε ελέγχου τη Eurostat. Και πολλά κράτη-μέλη απέρριψαν αυτόν τον κανονισμό γιατί δεν επιθυμούν το ρόλο αυτό να το διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω όμω η κρίση να μα δίδαξε ορισμένα πράγματα. Ε, η κρίση κατέδειξε την όλο και, μεγαλύτερη αλληλεξάρτησή μα. γιατί η κρίση αυτή οικονομική δεν είναι εθνικό ζήτημα. Μπορεί να έχει εθνικό χαρακτήρα, αλλά αφορά και το συλλογικό κοινοτικό συμφέρον. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε ενίσχυση του συντονισμού. Ο κύριο Άγερ, ο κύριο Βόμποτα, η κυρία Σαρνέ συμφωνούν ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη συντονισμένης ε, οικονομικής και δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής. Και Ευχαριστώ τον κύριο Σβόμποντα που μίλησε για φιλοδοξία και για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και όταν μιλούμε για τις δημοσιονομικές προοπτικές, ε, δεν θέλω να ενδώσουμε στον πειρασμό και να ενισχύσουμε το διακυβερνητικό σκέλος, γιατί η συνθήκη της Λισαβόνας ε, το αντίθετο δρόμο ακολουθεί, της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διάστασης και όχι της διακυβερνητικής. Α εκμεταλλευτούμε αυτή την κρίση για να ενισχύσουμε την Ευρώπη και να μην την αποδυναμώσουμε. Η κυρία Τεσσαρνέ μίλησε για το τη ρύθμιση στα χρηματοπιστωτικά θέματα. Είναι περίεργο, να μην πω ηρωνικό, ότι μετά από τέτοια αιτήματα και μετά από τέτοια ανάγκη, τα κράτη-μέλη ομόφωνα τελικά συμφώνησαν να περικόψουν τις φιλοδοξίες και να κόψουν τα φτερά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την έκθεση Τελαροζιέρ. Κάτι που δείχνει την ε, μεγάλη απόσταση που υπάρχει πολλές φορές και τη διαφορά μεταξύ των διακηρύξεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται τελικά. Ελπίζουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα μεταξύ λόγων και έργων και να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη συνοχή σε επίπεδο ευρωπαϊκής δράσης, γιατί πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη φιλοδοξία. Το μείζον πάντως ζήτημα εδώ είναι να αντιληφθούμε σωστά την αρχή της επικουρικότητας. Εγώ είμαι υπέρ της επικουρικότητας και συμφωνώ με τον κύριο Κίρκχοπ ότι είναι καλή η επικουρικότητα. Αλλά τι θα πει επικουρικότητα. Επικουρικότητα είναι να βρούμε το βέλτιστο επίπεδο για τη λήψη απόφασης. Η κρίση της εναέρειας κυκλοφορίας ε, δεν είναι περίεργο που συμβαίνει, γιατί είδα στο, διάβασα στον τύπο και όχι μόνο στο σκανδαλοθυρικό ή στον ευρωσκεπτιστικιστικό, διάβασα και σε σοβαρές εφημερίδες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραδέχεται τώρα ότι έλαβε και σφαλμένες αποφάσεις σε ό,τι αφορά την ακύρωση πτήσεων. Ε, αυτό πραγματικά είναι άνω ποταμών, γιατί αν υπάρχει ένας τομέας που αποτελεί αποκλειστική εθνική αρμοδιότητα, είναι ο τομέας των εναέριων μεταφορών. Η κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή λαμβάνει τη σχετική απόφαση. Και τώρα αυτοί που είναι κατά της ευρωπαϊκής δράσης αντιδρούν κατά της ε, αδράνη Ευρώπης. Μου πείτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φταίει που εξεράγει το ηφαίστειο στην Ισλανδία. Αυτό πραγματικά είναι ένα ποταμόν. Ας είμαστε σαφεί. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ευθυνών. Υπάρχει το εθνικό επίπεδο και το ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βρίσκουμε το καλύτερο επίπεδο για να αναλάβουμε δράση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνε της. Αλλά θα πρέπει να συμμαχίσουμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποσαφηνίσουμε τις ευρωπαϊκές ευθύνες από τις υπόλοιπες. Ή δεν θα έχουμε πάντα αυτό το αντανακλαστικό. Και φυσικά όταν σφίγγουν τα πράγματα, όταν έχουμε κρίσεις, είναι πολύ πιο εύκολο να ενδίδουμε σε δημαγωγικές ομιλίες και επιχειρήματα. Και πολλές φορές λένε ότι οι Βρυξέλλες φταίνε, το Στρασβούργο για κάτι που έγινε, ενώ στην ουσία αυτό αποτελεί εθνική αρμοδιότητα και ευθύνη. Επίσης θα πρέπει να πρετανεύσει και η κοινή λογική. Σε αυτό που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να επιφέρει προστιθέμενη αξία στις εθνικές δράσεις που είναι δημοκρατικές, γιατί πρόκειται για δημοκρατικές χώρες. Και το πρόγραμμα του 2020 επικεντρώνει την προσοχή μας στα ουσιώδη. Το ουσιώδες είναι η ανάπτυξη, αλλά όχι η ανάπτυξη ανεφόρων, ανάπτυξη πιο ε, δίκαιη, πιο φιλοπεριβαλλοντική, πιο αηφόρος, πιο ευφυής, στραμμένη προς το μέλλον. Χρειαζόμαστε νέες πηγές ανάπτυξη στην Ευρώπη. Έτσι μόνο θα αντιμετωπίσουμε το πιο σοβαρό πρόβλημα που θα εξετάσουμε το απόγευμα και που είναι η μάστιγα της ανεργίας και δι, της των νέων. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτή τη συμμαχία μεταξύ των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και φυσικά σε στενή συνεργασία και με τα κράτη-μέλη για να δουν οι πολίτες μας απτά αποτελέσματα. Και νομίζω ότι το πρόγραμμα αυτό είναι μια καλή βάση για το μέλλον. Και μετά τη συζήτηση νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκαρδιώθηκαν από τα ενθαρρυντικά σας σχόλια και θα φροντίσουμε να ανταπεξέλθουμε στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την απάντησή σας. Θα ήθελα να πω ότι σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στα θέματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μπορείτε να υπολογίζετε στην Συμμαχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών υποστηρίζει τις δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την προσέγγιση της για ανάληψη μεγαλύτερη ευθύνη ιδιαίτερα σε κρίσει. Γιατί τέτοιες κρίσεις δείχνουν τι επιτακτική ανάγκη υπάρχει για ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άλλωστε και οι δικέ μα αρμοδιότητε ενισχύθηκαν με τη συνθήκη τη Λισαβόνα και χαιρόμαστε γιατί πιστεύουμε ότι έτσι θα εξυπηρετήσουμε του Ευρωπαίου πολίτε. Να αναλάβουμε τι ευθύνε μα που είναι ενισχυμένε και να αξιοποιήσουμε τι δυνατότητε που μα δίνει η συνθήκη. Σα διαβεβαιώ, κύριε Πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα βρείτε σύμμαχο. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Υπουργό Λόπε Γκαρίντο για να μα εκφέρει και τη δική του γνώμη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να λάβω το λόγο απλά και μόνο για να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Πρόεδρο της ε, κύριο Μπαρόζο για αυτό το ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα που είναι ιδιαίτερα ευρωπαϊστικό και που μας παρουσίασε εδώ που βρίσκεται φυσικά σε απόλυτη συμφωνία με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής, Συμφωνία, της Ευρωπαϊκής Προεδρίας ε, αλλά και του τρίου των Προεδριών Ισπανίας, ε, Βελγίου, ε, Ουγγαρίας να πω ότι το Συμβούλιο συνεργάζεται στενά με την Κομισιόν αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο συγχαίρω για τις επικοδομητικές παρεμβάσεις υποστήριξης αυτού του νομοθετικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες. Όλοι γνωρίζουν ε, πως η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα η Επιτροπή Μπαρόζο 2 θα πρέπει θα έπρεπε μάλλον να αρχίσει να εργάζεται από την 1η Νοεμβρίου 2009, αλλά καθυστέρησε για ποικίλου λόγους ε, και ότι υπήρξε καθυστέρηση, έχει εργαστεί μέχρι τώρα ιδιαίτερα επικοδομητικά τους ε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπαρόζο και όλα τα μέλη της Επιτροπής, ε, αντιπροέδρους, ε, επιτρόπους. Πράγματι, αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που έχει καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά επίσης είχε μια θετική αντιμετώπιση και δράτω με τις ευκαιρίες ε, για να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια ακόμα φορά να μπορέσουμε σε αυτές τις ε, νομοθετικές πρωτοβουλίε ε, να εγκριθούν το συντομότερο δυνατόν έτσι ώστε να ανακτήσουμε τον χαμένο χρόνο στον οποίο αναφέρθηκα και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε την απόλυτη συνεργασία του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την απάντηση του Συμβουλίου και για την υποστήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μπαρόζο, και όλους τους αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους επιτρόπους για την παρουσία τους. Κάτι που δείχνει ε, τι σημασία και σπουδαιότητα δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μα χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Αυτά και ολοκληρώνεται η συζήτηση. Mr. President, thank you. Good to Sorry, I'm just looking for the for the. So colleagues, our next and last. Συνάδελφοι, το επόμενο και τελευταίο σημείο σήμερα διάταξη